Καθίστε παρακαλώ για να καθίσουμε, για να αρχίσουμε. Ευχαριστώ και καλώς ορίσατε στη συνεδρίαση. Σας ευχαριστούμε που ήρθατε σήμερα πέμπτη πρωί. Και το πρώτο θέμα είναι η έγκριση της ημερησίας διάταξης. Έχει υποβληθεί κάποιο αίτημα. Ε, συμφώνησαν οι συνεισηγητές για να αλλάξουμε τα σημεία 5 και 6. Να αναλογούν επομένως το 6 θα συζητηθεί πριν το σημείο 5. Έχετε κάποια αντίρρηση, επομένως με αυτή την αλλαγή να εγκρίνουμε την ημερησία διάταξη. Ωραία, σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε ανακοινώσει ε, Προέδρου. Ε, και επομένως τώρα προχωρούμε εις την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η πρώτη ψηφοφορία είναι το θέμα που αφορά τα σοφρονιστικά συστήματα και συνθήκες στις φυλακές. Η Μπάρμπαρα Ματέρα είναι η, η η οποία δεν παρίσταται. Επομένως δεν μπορεί να λάβει τον λόγο. Θέλει κάποιος άλλος τον λόγο. Γάλλους να προχωρήσουμε προς την ηλεκτρονική ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι? Έτοιμοι, ωραία. Και πάμε στην παράγραφο υπαριθμών 1 Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές ομόφωνη έγκριση από ό,τι φαίνεται. Πρώτη παράγραφος τροπολογία 8 χωριστή ψηφοφορία. Το πρώτο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά εγκρίνεται. Συμβαστική παριθμών 2. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο 14. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και πάμε τώρα στο 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική, όχι διορθώνει πρόεδρος 25 υπέρ κατά αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται. Για να δούμε το 25 υπέρ, κατά, αποχές. Εγκρίνεται. Μάλιστα. Ηλεκτρονική επαλήθευση για το 25. εγκρίνεται. 16. Ε, το 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται.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 αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, α, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, α, αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ, κατά, α, αποχές εγκρίνεται. Και τώρα με ηλεκτρονική ψηφοφορία όσον αφορά την τελική ψηφοφορία του σχεδίου γνωμοδοτήσεως. Ψηφίζουν. Πέρας. Εγκρίνεται 22 ψήφοι υπέρ. Σας ευχαριστώ πολύ και πάμε τώρα στη δεύτερη ψηφοφορία. Ε, σχετικά ε, με τον ε, διάλογο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. η πρόεδρος κανονικά ήταν η γνωμοδότρια στο συγκεκριμένο κείμενο. θα ξεκινήσουμε όμως με την ψηφοφορία. αρχικά ε, θα εξετάσουμε τα σημεία όπως βρίσκονται στην λίστα ψηφοφορίας ε, όσον αφορά τη στρατηγική για την ισότητα των φύλων υπερκατά αποχές εγκρίνεται ε, ισορροπία ε, στον συνδυασμό επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής ε, υπέρ, κατά, αποχές οπότε εγκρίνεται και τώρα όσον αφορά την έμφυλη βία η ψηφοφορία αυτή θα γίνει κατά τμήματα το ε, πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα όσον αφορά το τέταρτο σημείο, της ε, γυναίκες ε, στα διοικητικά συμβούλια και διαδικασία λήψης αποφάσεων, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται το συνταξιδοτικό χάσμα λογοφύλου υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται το ε, ανθρώπων υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται η συμμεταχείριση στην απασχόληση υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται το ε, κλείσιμο του ε, ψηφιακού χάσματος με βασταφύλλα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εδώ έχουμε μια ε, ψηφοφορία κατά τμήματα. Όσον αφορά το πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές. Το δεύτερο κομμάτι τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και το τελευταίο όσον αφορά την σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα υπέρ κατά εγκρίνεται. Οπότε κλείνουμε με την ηλεκτρονική ψηφοφορία και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο, στο σημείο 5, 6 μάλλον, ε, το οποίο μεταχειριστήκαμε ε, ως ε, νούμερο 5.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 Uh, Μπορούμε να αρχίσουμε και πάλι, διότι έχουμε αρκετά να συζητήσουμε σήμερα το πρωί. Ε, τώρα θα συζητήσουμε το σημείο 6 της ημερήσιας ε, διάταξης, ε, το οποίο αφορά την εφαρμογή της οδηγίας 2011-93 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κατομποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας στην προηγούμενη νομοθετική περίοδο η Επιτροπή ε, πρότεινε μια γνωμοδότηση ε, σχετικά με την καθορλόμηση της ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης ε, και παιδικής πορνογραφίας και είχαμε μια συμφωνία πλαίσιο του 2004 και τώρα, κάθε το 68 και τώρα θα έχουμε μια έκθεση από την πλευρά της ΛΥΜΠΕ θα αποφασίσαμε να έχουμε μια έκθεση εμείς που θα δοθεί στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ αποφασίσαμε να γίνει αυτό στις 16 Ιουνίου το οποίο όμως καθυστέρησε λόγω της καθυστέρησης της Κομισιόν Κομισιόν ε, για την έκδοση της έκθεσής της σχετικά με την εφαρμογή της ε, ε, οδηγίας. Θεωρούμε ότι το ζήτημα του φίλου θα πρέπει να συμπεριληφθεί για την προστασία της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών. Θα δώσω όμως το λόγο τώρα στην γνωμοδότρια κυρία Μούντι. As you rightly said, uh, the, our opinion to the LIBE Committee on uh, how the directive has been working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 Αυτό ίσως ε, δημιουργεί περισσότερες ε, διαφωνίες. Το θέμα είναι πώς κανείς το βγάζει από το ίντερνετ και πώς το ε, απαλήφει εντελώς. Και εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Και τέλος, η παρέμβαση, η πρόληψη και η κατάρτιση. Πώς θα παρέμβουμε έναντι αυτών που χρηματοδοτούν. Είναι δύσκολο ούτως ή άλλως. Συγγνώμη, ε, η παρέμβαση έναντι ε, των ε, ατόμων που έχουν καταδικαστεί για κάποια τέτοια αδικήματα και πώς θα τους βοηθήσουμε να μην ε, διαπράξουν και άλλα ε, τέτοια, τέτοιου τύπου αδικήματα. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κοράτσα Μπίλτ. Ευχαριστώ Κλέα. Εργαστήκαμε πολύ καλά μαζί και βλέπω ότι συμμετείχες και στην ακρόαση που κάναμε για το θέμα αυτό στη Λίμπε. Είμαι η συγγήτρια στη Λίμπε για την οδηγία αυτή για την εφαρμογή και αναθεώρηση. Δυστυχώς υπάρχει μια ε, πολύ έντονη διάσταση φύλου. Πλήττονται πολύ περισσότερο τα κορίτσια. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ιδρύματος που παρακολουθεί το ίντερνετ, Internet Watch Foundation, η Ευρώπη έχει ε, το υψηλότερο ποσοστό τέτοιου ποσοστού τέτοιου περιεχομένου κακοποίησης και είναι 60% της ε, συνολικής τέτοιου τύπου συμπεριφοράς και έχει υπάρξει και τεράστια αύξηση, 90%. Επίσης, αναφέρει η έκθεση αυτή ότι αυξάνεται η δική μας ε, η παρουσία τέτοιων φαινομένων στην Ευρώπη ενώ στη Βόρεια Αμερική μειώνεται και τα κορίτσια κυρίως είναι θύματα και οι περισσότερες επαφές που, γίνεται, που γίνονται με τέτοια ευάλωτα άτομα γίνονται μέσω του ίντερνετ. Συμφωνώ πολύ με τη γνωμοδότησή σας. Να αναφέρω όμως μερικά θέματα που θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν στην έκθεση στη Λίμπε Και εσείς ε, παραλαμβάνετε ε, την, πορνογρα... την εκδικητική πορνογραφία νέου τύπου ε, αδικήματα είναι αυτά, εγκλήματα τα οποία διαπράττονται Πρέπει να δούμε δηλαδή τι νέου είδους εγκλήματα διαπράττονται από τότε που εγκλήθηκε η οδηγία και σωστά τα αναφέρεις Κλέα, αυτή την εκδικητική φωνογραφία που έχει κατόπιν ως συνέπεια κάποια κορίτσια να αυτοκτονούν στο ίντερνετ, στο facebook γιατί δεν μπορούν να ανεχθούν τον αριθμό από εικόνες ε, ή άλλο περιεχόμενο από τη σεξουαλική τους ζωή που χωρίς τη δική τους έγκριση ανεβαίνουν στο ίντερνετ. Επίσης υπάρχει πολύ περισσότερο το grooming, η προετοιμασία δηλαδή ε, ατόμων για να συμμετάσχουν ε, κατόπιν σε τέτοιες διαδικασίες και επίσης εκβιασμός. Επίσης, συμφωνώ με αυτά που λέτε για τον κίνδυνο ακριβώς αυτής της διάδοσης ε, περιεχομένου και πώς πρέπει να καταρτήσουμε τους εκπαιδευτικούς, ε, τους κοινωνικούς λειτουργούς, αυτούς που ασχολούνται με το, τους εργαζόμενους στο δικαστικό σύστημα. Πρέπει ακριβώς μέσω αυτής της δικαστικής διαδικασίας να αποφύγουμε επιπλέον βλάβη ε, προς τα θύματα, πώς ε, κάνουμε τις ερωτήσεις, πώς ε, τις ενθαρρύνουμε, ενθαρρύνουμε τα θύματα γενικά να αναφέρουν τα προβλήματά τους χωρίς να χρειάζεται να πούν 20 φορές το ίδιο πρόβλημα σε διάφορους αστυνομικούς και δικαστικούς. Πρέπει να προστατεύσουμε το θύμα ούτως ώστε να αποδοθεί πραγματικά δικαιοσύνη. Και επίσης πρέπει να ενισχύσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών. Η Ευρωπόλ κάνει θαυμάσια δουλειά επ' αυτού. Πριν από δύο εβδομάδες κατάφεραν να διαλύσουν ένα τέτοιο δίκτυο στην Ανατολική Ευρώπη. Και το Eurojust έχει ε, ένα τμήμα που εργάζεται ακριβώς για αυτήν την επιγραμμική κακοποίηση παιδιών. Πρέπει να έχουμε εθνικά μητρώα και υπηρεσίες προστασίας των παιδιών. Είναι πολύ σημαντικό να μας δώσει ταχαίως ε, πολύ περισσότερη πληροφόρηση κομισιών. Τώρα πήραμε μόνο αυτή τη μελέτη για το πώς εφαρμόζουν την οδηγία τα κράτη-μέλη. Βλέπουμε ήδη ότι υπάρχουν ε, πολύ σοβαρές ανεπάρκειες σε πολλά κράτη-μέλη αλλά δεν έχουμε επαρκή πληροφόρηση. Θα ήθελα να εστιάσω στο θέμα της εφαρμογής. Υπάρχουν και άλλα θέματα που είναι επίσης σημαντικά για την πρόληψη. Το βλέπουμε ιδίως με βάλω τα παιδιά όπως ε, ασυνόδευτα παιδιά μεταναστατικού, μεταναστευτικού, μεταναστευτικής προέλευσης Πρέπει να ενημερώσουμε και τους κηδεμόνες, τις οικογένειες τις οποίες, ε, οι οποίες ασχολούνται με αυτά τα παιδιά, που έχουν αναλάβει δηλαδή αυτά τα παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία και θα κάνω την μπορώ τόσο ώστε στη Λίμπε να συμπεριληφθεί στην έκθεσή μας η γνώμη σας. Ευχαριστώ. Η κυρία Ζιντζινιάμσκα. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Πολύ καλό κείμενο, χαίρομαι για τη συνεργασία. Δεν έχω και πολλά να πω, γιατί πολύ σωστά παρουσιάσετε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε με αυτά τα νέα φαινόμενα μέσω της χρήσης ε, των κοινωνικών μέσων. Θα ήθελα ίσως να εμπλουτίσω λίγο το κείμενό σας με παρατηρήσεις για τις γυναίκες και τα παιδιά από την κοινότητα Ρωμά που είναι πολύ ευάλωτη στην Σλοβακία και επίσης ε, παιδιά με αναπηρίες και αυτά είναι πολύ ευάλωτα δεύτερη παρατήρηση Πώς θα συνειδητοποιήσουν και οι γονείς περί τίνος ε, πρόκειται πολύ συχνά εμφανίζονται γυμνές φωτογραφίες παιδιών, ακόμη και βρεφών, τα οποία, οι οποίες φωτογραφίες και περιεχόμενο κατόπιν αναμεταδίδονται από αυτούς τους εγκληματίες. Αυτήν την συμπεριφορά πρέπει να την ε, καταπολεμήσουμε, αυτά τα φαινόμενα. Και αυτά που είπατε και εσείς και η κυρία Κοράτσα Μπίλτ για την εκδικητική πορνογραφία. Και αυτό νέο φαινόμενο. Πρέπει να το συζητήσουμε και χαίρομαι που το συμπεριλάβατε στην γνωμοδότησή σας για έξι χρόνια στην Σλοβακία ήμουν μέλος ενός εποπτικού συμβουλίου ραδιοτηλεοπτικών μέσων και Παρακολουθούσαμε καθημερινά επί πολλέ ώρε προγράμματα, ε, άρα αυτό, τέτοιου περιεχομένου. Η προγραφία λοιπόν δεν έχει όρια, πρέπει να συνεργαστούμε όλοι. Ευχαριστώ πολύ, χαίρομαι για την ε, συνεργασία που θα έχουμε. Ευχαριστώ κυρία Μπεθέρα. Εγώ ευχαριστώ πρόεδρε και θέλω να ευχαριστήσω όμως και την κυρία Μούντι, αλλά και την κυρία Κόρατσα Μπίλτ για αυτή την κοινή προσπάθεια όσον αφορά την εφαρμοστική αυτή έκθεση. Νομίζω ότι τελικά α, το πιο πολύτιμο που μπορούμε εμείς να συνεισφέρουμε σε αυτή την προσπάθεια, πώς να σας το πω, είναι να προσπαθήσουμε να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, να μπορέσουμε να συντονιστούμε με την ταχύτητα με την οποία οι εγκληματίες ε, χρησιμοποιούν και κατά χρόνια εκμεταλλεύονται τα παιδιά από πλευρά σεξουαλική όσον αφορά αυτή την παιδική πορνογραφία. Αυτοί ε, προσαρμόζονται πάρα πολύ γρήγορα ε, και βλέπουν που υπάρχουν οι ευκαιρίε τόσο ώστε να κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν και επίση ε, θα πρέπει να μπορέσουμε να ενημερωθούμε όσον αφορά τα νέα μέσα που εκείνοι χρησιμοποιούν και κυρίως να μην παρασυρώμαστε ε, όσον αφορά την πρόληψη και να δούμε πού επεκτείνεται, πού διευρύνεται ε, αυτή η δραστηριότητα της παιδικής ε, πορνογραφίας. Επίσης ε, να λάβουμε υπόψη τι γίνεται στις χώρες μας από τις διοκτικές αρχές, στη ΔΕ η Ισπανία υπάρχει πάρα πολύ καλός συντονισμός μεταξύ αυτών των ε, αρχών και των αντιστοίχων Ευρωπαίων ομολόγων τους. Οπότε όταν είναι τόση αποτελεσματικότητα αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε έναν ολόκληρο στρατό από εγκληματίες αυτοί οι οποίοι είναι προσανατολισμένοι ε, σαφώς προς το την ε, κακοποίηση, την σεξουαλική, την εκμετάλλευση των ανηλίκων μέσα σε αυτό το, το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον στο οποίο ζούμε έχουν όλα τα σχετικά μέσα και εργαλεία. Επομένως θέλουμε να βοηθήσουμε σε αυτή την έκθεση και να αναγνωρίσει η κοινωνία σαφώς τις επιπτώσεις της πορνογραφίας και επίσης τις σεξουαλικές επιθέσεις. Να αναγνωριστεί ότι υπάρχει μια τέτοια σχέση και ήδη αυτό έχει αναγνωριστεί σε κάποιες χώρες όπως την Νορβηγία. Δεν είναι δυνατόν επομένως να υποτιμήσουμε την επίπτωση αυτή της πορνογραφίας ούτε να την αποσυνδέσουμε με το άλλο φαινόμενο δηλαδή των σεξουαλικών κακοποίησεων και επιθέσεων και ποιήσεις εντάξει να μην ποινικοποιούμε εκ των ε, προτέρων αλλά θα πρέπει επίσης να δούμε ποιοι είναι οι πιο ευάλωτοι όσον αφορά την επιμέλεια των ε, ανηλίκων και στο σύνολό της η κοινωνία έχει υποχρέωση να φροντίσει, να προσέξει τους ανηλίκους. Αυτό είναι κοινή ευθύνη και επίσης θα πρέπει να είμαστε εξοπλισμένοι με μια σταθερή ε, προσπάθεια πρόληψης. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να τίνουμε ευήκοους προς αυτό που έχουν να πούν σε μας οι ανήλικοι φυσικά και διαφέρουν πολύ ένομε τάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψη το τι λένε οι ανήλικοι. Πέραν της ψυχολογικής υποστήριξης και ανακούφισης κάθε φορά της έρευνας αλλά να ακούμε τα παιδιά και εκεί θα πρέπει να υπάρχει κάποιο είδου ε, εναρμόνιση του τι καταθέτουν τα παιδιά, το πώς αυτό λαμβάνεται υπόψη, υπό ποιου όρου γίνεται τούτο. Ε, ευχαριστώ, εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, η επόμενη μιλήτρια, η κυρία Αγιούτο Πρόεδρος, παρακαλώ να είμαστε σύντομοι, γιατί έχουμε και άλλη συζήτηση και άλλη έκθεση και πρέπει 10 η ώρα να αρχίσει η ακρόαση. Σύντομα παρακαλώ λέει η πρόεδρος. Ναι, ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, λέει η κυρία Αγιούτο και ευχαριστώ την εισηγήτρια. Ναι, όλα αυτά τα οποία είπατε, για μια που βρισκόμαστε τώρα ενώπιον αυτού του είδους μορφής βίας κατά των γυναικών. Αλλά η ε, ε, δυνάμια αυτό ε, στρέφεται κατά όλων. Λίγα γνωρίζουμε ακόμα. Και επίση μέσον είναι το ίντερνετ και το θέμα είναι αν υπάρχει συνένεση ε, ε, πολλές φορές ε, κάποιοι κρύβονται πίσω από μία οθόνη ε, και οπότε έτσι κάποιος καθίσταται θύμα αυτής της προσπάθειας και δεν έχουμε επαρκή μέσα για την προστασία των πάντων και ακόμη περισσότερο για να προστατεύσουμε τους ανήλικους, που πολύ νέους, πολύ μικρούς, που ακόμα δεν έχουν την οριμότητα να προστατεύσουν εαυτόν. Οπότε οπωσδήποτε θα πρέπει να προβλέπονται ποινές κατά αυτών που χρησιμοποιούν πορνογραφικό υλικό και, ό, και ό,τι συλλέγουν σαν φωτογραφίες χωρίς συνένεση. Πολλές φορές οι νέοι με τη συνένεσή τους ε, ανεβάζουν στο διαδίκτυο υλικό που αφορά ιδιωτικέ ε, προσωπικές στιγμές. Όμως δεν ξέρουν τι κίνδυνοι ελοχεύουν από τέτοιες ενέργειες. Το κάνουν αυτό από ανοριμότητα, από έλλειψη επίγνωσης των συνεπειών και όσον αφορά τον σεξουαλικό τουρισμό. Αυτό είναι μια άλλη πληγή και εδώ επίσης το, το θέμα σηκώνει τιμωρία γιατί έχουμε πολλούς Ευρωπαίους το κάνουν αυτό αλλά υπάρχουν επίσης και κάποιες γραφεία που διοργανώνουν τέτοια ταξίδια τουριστικά εντό εισαγωγικών. Και ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος και δίνω το λόγο στην κυρία Βόρντ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ε, πολύ καλό το ότι βλέπω τη συναδελφό μου κυρία Μούντι να εργάζεται πάνω σε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση. Ε, ε, και συγκεκριμένα γνωρίζοντας ε, ότι η συνεργασία, η διασυνοριακή συνεργασία είναι ένας πολύ σημαντικός ε, τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο φαινόμενο. Ως Βρετανοί Ευρωβουλευτές γνωρίζουμε ότι υπάρχει πολύ σοβαρός κίνδυνος εξαιτίας του Brexit για την ασφάλεια των παιδιών στο online περιβάλλον. Είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό. Βρίσκομαι επίσης στην Επιτροπή Κουλτ ε, και ε, όποτε εργάζομαι σε εκθέσεις εκεί πέρα, τότε φροντίζω αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι η σεξουαλική εκπαίδευση. Ε, θα πρέπει οι νέοι να έχουν εκπαιδευτεί και να σέβονται ο ένας τον άλλον, να γνωρίζουν ποιες είναι οι σωστές και υγιείς σχέσεις και το πώς να συμπεριφέρονται ο ένας τον άλλον και πώς να περιμένουν ότι θα τους συμπεριφέρονται οι άλλοι. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουμε το συγκεκριμένο ζήτημα πιο σοβαρά. Είναι καλό το γεγονός ότι ε, μιλήσαμε για τα δικαιώματα των παιδιών και ακούσαμε και τις απόψεις των παιδιών πάνω σε αυτό. Έχουμε ε, εργαστεί πάνω στην ε, ομάδα για τα δικαιώματα των παιδιών και όσον αφορά τη θυματοποίηση και οποιαδήποτε μορφή βίας κατά των παιδιών είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό το οποίο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εκ μέρους μας στην ομάδα αυτή. Και ε, επίσης θέλω να προσθέσω ότι και τα ΜΜΕ παίζουν ένα πολύ σοβαρό ρόλο σε αυτό. Τα μέσα αλλά και οι διαφημίσεις έχουν δημιουργήσει ένα ε, κλίμα ε, μέσα στο οποίο τα κορίτσια και τα παιδιά γενικότερα ε, βλέπουν ε, το ρόλο τους ε, ως αρκετά σεξουαλικό. Αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο και υποστηρίζει ένα περιβάλλον στο οποίο η βία κατά των γυναικών και των παιδιών αποτελεί κομμάτι της κοινωνίας μας και αυτό είναι ιδιαίτερα στενάχωρο τη σήμερα εποχή. Όσο πιο γρήγορα λοιπόν τα κράτη-μέλη εγκρίνουν την σύμβαση της Κωνσταντινούπολης τόσο το καλύτερο. Τα κράτη, οι γυναίκες δεν είναι ορατέ ε, στην ε, κοινωνία μας με αποτέλεσμα κατά συνέπεια στη συνέχεια ε, οι γυναίκες να αντιμετωπίζονται ως πράγματα. Αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα και δεν θα πρέπει να το εξετάσουμε ως κάτι διαφορετικό από άλλα σημεία της κοινωνίας. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα περάσουμε στην κυρία Χιούμανες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια, την κυρία Μούντι, και την Αναμαρία βέβαια που χαίρει μεγάλης εκτίμησης γιατί εδώ και πολύ, πολλά χρόνια εδώ στο σώμα μας ε, αγωνίζεται για τα δικαιώματα των ε, παιδιών. Οπότε είναι πολύ θετικό που είναι και στη Λίμπε και στη ΦΑΜ γιατί οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει το θέμα αυτό με την ε, γνωστή της αφοσίωση. Πολλοί από εσά μιλήσατε για την πορνογραφία να θυμίσω ότι όταν ξεκινήσαμε αυτήν την έκθεση το 2011 συζητούσαμε για το ίντερνετ και την φωτογραφία και την πορνογραφία, αλλά αυτή η έκθεση μιλάει και για την κακοποίηση των παιδιών που δεν γίνεται μόνο μέσω του ίντερνετ αν και είναι και πολύ σημαντικό αυτό δεν χρειάζεται να το επαναλάβω η έκθεση λοιπόν ε, θα μας βοηθήσει να δώσουμε ορατότητα στα θέματα αυτά. Το πρόβλημα που υπάρχει με την κακοποίηση των παιδιών είναι ότι τα παιδιά δεν μπορούν να εκφράσουν το πρόβλημά τους. Είναι πολύ δύσκολο να εκφράσουν τα παιδιά. Αυτό μας λέει η αστυνομία. Ερευνάει η αστυνομία, αλλά δεν υπάρχουν καταγγελίες. Γιατί? Γιατί συνήθως ε, συμβαίνουν αυτά σε περιορισμένα, σε κλειστά περιβάλλοντα, όπω τα σχολεία και η οικογένεια και κανεί δεν ξέρει. Αυτά όσον αφορά την Ευρώπη. Δεν μιλάμε για τη διακίνηση παιδιών κτλ. ή αυτά που συμβαίνουν σε άλλες ε, περιοχές. Δεν μιλάμε για αυτά που ε, δυστυχώς παθαίνουν ε, τα κορίτσια μετανάστες κτλ. Όχι. Μιλάμε για τα άλλα φαινόμενα. Χρειαζόμαστε στοιχεία. Πρέπει να δούμε πού προκύπτουν αυτά, πού υπάρχουν περισσότερα τέτοια φαινόμενα και να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά. Να μπορεί δηλαδή και η αστυνομία να παρέμβει. Επειδή δεν υπάρχει πολύς ε, χρόνος, να σταματήσω τώρα. Ευχαριστώ. Ήταν η τελευταία ομιλήτρια που ζήτησε το λόγο και τώρα ε, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να σας πω ε, το χρονοδιάγραμμα. Η ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών είναι στις 18 ε, Μαΐου, στη 1 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία στη ΦΕΜ θα γίνει στις 20 Ιουνίου, ενώ στις 7 Σεπτεμβρίου θα γίνει η ψηφοφορία από την πλευρά της ΕΜΠΛ. Θα ήθελα να προσθέσει κάτι η Κομισιόν. Ναι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Μούντι για την ε, συγκεκριμένη ε, γνωμοδότηση και ακολουθεί ε, τα ευρήματα τα οποία έχουμε τονίσει στην έκθεση της Κομισιόν που δημοσιεύθηκε πέρσι το Δεκέμβριο. Η Κομισιόν θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τα κράτη-μέλη για να διασφαλίσει την πλήρη εφαρμογή της οδηγίας και συγκεκριμένα όσον αφορά τα ζητήματα τα οποία αναφέρθηκαν στην γνωμοδότηση όπως είναι το ζήτημα της πρόληψης αλλά και την πληροφόρηση των κρατών μελών, την καταπολέμηση ε, του σεξουαλικού τουρισμού ε, καθώς επίσης ε, και την εκπαίδευση όσων εργάζονται με παιδιά αλλά και την ενίσχυση όσων προσπαθούν να καταπολεμήσουν το συγκεκριμένο φαινόμενο. Σας ευχαριστώ πολύ. Λέει η Πρόεδρος, Κλέρ, θα ήθελες κλείνοντας να προσθέσει κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για όλες σας τις συνεισφορές, θα τις λάβω υπόψη μου. Ο σκοπός αυτής της γνωμοδότησης είναι να διασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ε, μία ε, ισχυρή προσθήκη στην ε, έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ διότι τα αποτελέσματα του έργου που κάνουμε ε, είναι πολύ σημαντικά και είναι ε, ζωτική σημασίας ε, να τα συμπεριλάβουμε και να έχουμε μια σταθερή θέση πάνω σε αυτό. Θα συνεργαστώ με τους συναδέλφους. Καλωσορίζω το έργο της Άννα Μαρία πάνω σε αυτό και θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση με τις τρομολογίες. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε Κλέρ και ε, περιμένουμε με τιμωμονησία την ε, συζήτηση πάνω στο συγκεκριμένο θέμα. Και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 5. Ε, η συντάκτρια της γνωμοδότησης δεν βρίσκεται εδώ. πιστεύω η κυρία Χιούμανες θα μας παρουσιάσει το συγκεκριμένο θέμα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να μιλήσω αντί της κυρίας Λεγκρίπ, που είναι η συγγήτρια αυτή τη γνωμοδότηση όσον αφορά την εντολή για τον τριμερή διάλογο. Κυρία Λεγκρίπ, δυστυχώ δεν μπόρεσε σήμερα να παραστεί, οπότε σα ζητεί συγγνώμη για αυτό το λόγο και Πρόκειται για σχέδιο γνωμοδότηση, το οποίο έχει σκοπό τόσο ώστε να απευθυνθούμε στην Επιτροπή των Προπολογισμών σε σχέση με την κατάρτιση του προπολογισμού της ε, χρήσης του 2018 τόσο ώστε να καλυφθούν κάποια ε, βασικά σημεία τα οποία είναι πάρα πολύ ε, σημαντικά για τη δική μας Επιτροπή. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό τα ιδιωμή των γυναικών αλλά και των δύο φύλων να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό και κυρίως όσον αφορά την ορθή υλοποίηση κάποιων προγραμμάτων όπως το πρόγραμμα Δάφνη, το οποίο θα πρέπει να θεωρηθεί πάρα πολύ σημαντικό για αυτόν τον επόμενο προπολογισμό. Στο σχέδιο γνωμοδότηση η κυρία Λεγκρίπ τονίζει κυρίως το ότι θα πρέπει να προαχθεί η υπόθεση της ισότητας των δύο φύλων, θα πρέπει να καταπολεμηθούν δυσμενείς διακρίσεις και επίσης ότι θα πρέπει να χειροφετηθούν οι γυναίκες σε όλα τα επίπεδα. Επίσης έχει τονίσει το πόσο κρίσιμος είναι ο ρόλος του να καλυφθεί η ισότητα των ε, φύλων από την πολιτική μας, από τα προγράμματα όπως το ορίζουν 2020 και αυτά βοηθούν στην επίτευξη των ελόγων στόχων. Η κυρία Λεγκρίπ επίσης συστήνει στο ότι θα πρέπει να υλοποιηθεί αυτή η ένταξη και κάλυψη από τον προπολογισμό της όντας των φίλων. Είναι πολύ σημαντικό ότι η δική μας Επιτροπή επίσης θέλει να υπάρχει συγκεκριμένα ε, η υπόθεση μας αυτή για τον προεκλογισμό του 2018 και με αυτή την κάλυψη των προπολογισμών θα μπορούμε να έχουμε κάποια προγράμματα και αυτό θα γίνεται με τρόπο που θα γίνεται από διαφάνεια και αποτελεσματικότητα και να υπάρξει επίση και παρική προοικοδότηση. Επίση, τονίζεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και χρειάζονται οι γυναίκε να εμπλακούν περισσότερο, να χειραφετηθούν όσον αφορά τα τη ευρωπαϊκή οικονομία και ιδίω οι γυναίκε να συμμετάσχουν στην ψηφιακή επανάσταση και ε, στις τεχνολογίες ε, πληροφορίας και επικοινωνίας και αυτό που το πετύχουμε ε, αν εμπλακούν οι νέες γυναίκες στις θετικές επιστήμες, τεχνολογία κλπ. Οπότε έτσι θα υπάρξει περισσότερη συνειδητοποίηση του τι ευκαιρίες προσφέρουν αυτοί οι τομείς, θετικών επιστήμων δηλαδή κλπ. Και πληροφορίας οπότε μπορεί το Κοινοβουλίο να βοηθήσει για τέτοιου είδους δράσεις και το τονίζει αυτά στο κείμενο της η κυρία Λεγκρυπ. Τέλος, θέλει να υπενθυμίσει ότι θα πρέπει να υπάρξει οικονομική υποστήριξη μέσω του προβλησμού της χρήσης του 2018 και έτσι αυτό μπορεί να το κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης θα πρέπει να υπάρχουν δεδομένα που χρειάζονται όσον αφορά την ισότητα των φίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα δεδομένα και να δούμε πώ θα έχουμε καινοτόμε και αποτελεσματικέ πολιτικέ για να βελτιώσουμε την κατάσταση ισότητα των φίλων και την υπόθεση τη χειραφέτηση του. Το θέμα αυτό θα συζητηθεί 8 Ιουνίου και για τις τροπολογίες έχουμε προθεσμία μάλλον 16 Πέμπτου το μεσημέρι και θα γίνει συζήτηση των τροπολογιών κατόπιν στην Επιτροπή Προπολογισμών θα... Όχι, 8 Ιουνίου θα γίνει η ψηφιστική μας Επιτροπή και 19 ή 20 Ιουνίου στην Επιτροπή των προπολογισμών και στην Ολομέλεια μάλλον 6 Ιουλίου. Τίποτα άλλο. Η ιδέα για κυρία Λεγκρή προβλέπει στην υπεραιτέρω συνεργασία με τους συναδέλφους και σας ευχαριστούμε. Θέλει το λόγο κάποιος από τους κοιόδης εισηγητές. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την Κωνσταντζ Λεγκρίπ για το σχέδιο γνωμοδότησης όσον αφορά τον προπολογισμό. Αυτό είναι καλή ευκαιρία για συζήτηση. Εμεί οι πράσινοι θα κατεβάσουμε κάποιε τροπολογίε, ιδίω για κάποια διατύπωση, ιδίω εκεί που λέτε για το πώ θα πρέπει να ενταχθεί στον προπολογισμό, η ισότητα των φύλων και όμω θέλουμε να υπάρξει υλοποίηση είναι υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το mainstream της ισότητας των φίλων. Αυτό θα να τονίσουμε, γιατί καμιά φορά είναι απογοητευτικό ότι δεν τα εφαρμόζουν αυτά τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Τώρα, όσον αφορά το πρόγραμμα Δάφνη, όσον αφορά την καταπολέμηση τη βία κατά των γυναικών, και εδώ θέλουμε να είναι ε, πιο δυναμική η διατύπωση και επίση χρειάζονται περισσότερα κονδύλια και αυτό να καταστεί προτεραιότητα και χρειάζονται χρήματα από τον προπολογισμό για ασφάλεια. Θεωρούμε ότι η ατομική ασφάλεια των γυναικών είναι το ίδιο σημαντική όπως και η συλλογική ασφάλεια της κοινωνίας. Επίσης θέλουμε μια πιο δυναμική διατύπωση όσον αφορά την ανάπτυξη που θέλουμε να είναι βιώσιμη και όσον αφορά την αναδιανομή του πλούτου και αξιοπρεπή απασχόληση, όχι απλώς δουλειές να είναι αξιοπρεπεί αυτέ όσον αφορά την επαγγελματικό βίο. Και εδώ έχει σημασία ο προπολογισμό και επίση κάποια πιλωτικά προγράμματα για το mainstream τη όντα των φύλων και υπάρχει το πρόγραμμα εκείνο το οποίο λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν κάποια προγράμματα για τα θεσμικά όργανα αφορά αυτό μισό εκατομμύριο λέμε άρα θέλουμε να υπάρξει ένα τέτοιο κονδύλιο και τέλος καταβάζουμε κάποιε τροπολογίε για το πόσο σημαντική είναι η επενδυτική πολιτική στα πλαίσια τη πολιτική συνοχή για τα διαρθρωτικά ταμεία και επίση να κάνουν κάποιες ε, δαπάνες σχετικά. Και πω βλέπουμε στην συνεργασία με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Θέλει κανένα άλλο μέλο τη επιτροπή μα να πάρει το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ωραία. Κυρία Χιμένη, θέλετε να συνοψίσετε τη συζήτηση. Ναι, να απαντήσω. Φυσικά συμφωνώ. Πρέπει να υποβληθούν τροπολογίες για το mainstreaming φύλου. Βεβαίως. Δεν πρέπει να είναι μόνο λόγια πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη δέσμευση. Βεβαίως δεν ε, είμαι εισηγήτρια, αλλά είμαι εδώ και πολύ καιρό, πολλά χρόνια, μέλος αυτής της Επιτροπής, αλλά και της ΛΥΜΠΕ βεβαίως. Πρέπει να είναι προτεραιότητα να υπάρξει περισσότερη χρηματοδότηση για την καταπολέμηση της βίας με βάση το φύλλο. Καλό λοιπόν είναι να υποβληθούν αυτές οι τροπολογίες και μετά θα συζητήσουμε και το θέμα των δικαιωμάτων των θυμάτων που περιέχει πολλά για την βία λογοφύλου και για την προστασία των θυμάτων αυτού του είδους βίας. Είναι λοιπόν πολύ καλή ευκαιρία να εργαστούμε για το θέμα αυτό. Φυσικά πρέπει να προστατεύσουμε και να βοηθήσουμε όλα τα θύματα διακίνησης, τρομοκρατίας, οργανωμένου εγκλήματος, αλλά βεβαίως πρέπει να αναφερθούμε ιδιαίτερα στις γυναίκες που είναι θύματα βίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, υπενθυμίζω Προθεσμία για τροπολογίες 16 Μαΐου μεσημέρι 12, ψηφοφορία στην Επιτροπή 8 Ιουνίου, στην Μπάτζ 19 ή 20 Ιουνίου, στην Ολομέλεια στην 3, 3 με 6 Ιουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήσασταν και τόσο σύντομοι. Έχουμε ένα πεντάλεπτο πριν την έναρξη της ακρόασης, ένα σύντομο διάλειμμα παρακαλώ να είστε πίσω στις 10 γιατί πρέπει να ξεκινήσουμε ακριβώς στις 10.